την εφαρμογή και την επιλογή τη οδηγία 2059 ΕΚ για ε, τι αθέμενε εμπορικέ πρακτικέ των επιχειρήσεων προ του καταναλωτέ στην εσωτερική αγορά και τη οδηγία 2006-114 για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση. Ευθύνη τη βουλευτού κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ, στην οποία δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Βουλευτά, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν να, να σχολιάσω την έκθεσή μου, θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι πιστεύω ότι εμείς με την απόφασή μας ε, για τις εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας τα κάναμε λίγο θάλασσα. Τώρα που βλέπω πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις για αυτές τις εκθέσεις πρωτοβουλίας χωρίς συζήτηση, χωρίς ε, ε, διάλογο Νομίζω ότι πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε λίγο τις αποφάσεις μας. Τέλος πάντων για την έκθεσή μου τώρα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους με τους οποίους συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία ε, που μας βοήθησε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς έβαλε το θέμα την έκθεσή μου αρκετά ε, νωρί, στην ημερήση ημερήσια διάταξη, το πρόγραμμα εργασιών της ε, συνειδητά για να μπορέσουμε να ε, ε, δούμε ε, τα πώς προχωρούν τα πράγματα πως ήταν το 2007 από εκεί και πέρα βέβαια δεν έχουν γίνει δεν έχουν αλλάξει τρομακτικά τα πράγματα αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τρία κράτη-μέλη που δεν κατάφεραν να τηρήσουν αν θέλετε κάποιες προθεσμίες και εδώ μιλάμε για ιδρυτικά κράτη-μέλη δεν μιλάμε για νέα κράτη-μέλη που δεν γνωρίζουν το κοινοτικό δίκαιο τέλο πάντων τρία κράτη-μέλη δεν έχουν εντάξει εθνικές τους νομοθεσίες ακόμη τη, τη οδηγία υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κύρωσης και υπάρχουν όμως και προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με άλλα λόγια με δυο λόγια μάλλον κακή εφαρμογή μάλλον ελλειπής εφαρμογή της οδηγίας από εκεί και πέρα υπάρχουν κράτη-μέλη, υπάρχει η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστρία που εφαρμόζει 100% την οδηγία αυτή και ίσως πάει και παραπέρα. Εμείς η οδηγία αυτή εγκρίθηκε για να βελτιώσει τα πράγματα για να προστατεύσει τους πολίτες, τους καταναλωτές από ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές και για τις μικρές, ε, ιδιαίτερα για τις μικρές επι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ότι αυτό πρέπει να ε, το λάβει ιδιαίτερα υπόψη η Επίτροπος διότι τελικά πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τα ίδια προβλήματα με τους καταναλωτές έτσι δεν είναι στη μεριά των μεγάλων επιχειρήσεων που είναι απέναντι στον καταναλωτή τέλος πάντων ε, ποιες είναι οι αθέμητες πρακτικές ξέρουμε ότι συμβαίνουν πολλά στην Ευρώπη ελαχία λαχεία ε, αυτά που γίνονται με τους ταχυδρομικούς κώδικες ε, στοιχήματα κτλ ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έρθει να έχει στενότερη επαφή με τις ε, εθνικές ε, αρμόδιες αρχές και ε, να παρακολουθείς και το θέμα αυτών των μαύρων καταλόγων, των μαύρων ληστών που υπάρχουν. Ε, γενικότερα ίσως ισχύει αυτό που θα πω τώρα αλλά νομίζω ότι και εδώ πρέπει να το πούμε ότι χρειάζεται συνεργασία χρειάζεται συνεργασία και με τους πολίτες και με τους θεσμούς και με τα όργανα της κοινότητας και οι βουλευτές μας θα πρέπει να παρακολουθούν τις χώρες τους. Αν το είχαν κάνει θα εφαρμοζόταν καλύτερα οι οδηγίες αυτές. Η κυρία Βασιλείου. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Βάιλερ για την έκθεσή της την οποία θα την μελετήσουμε ενδελεχώς στην Κομισιόν. Ευχαριστώ όμως και για τα σχόλια που έκανε σχετικά με τη διαδικασία. Η Κομισιόν συμφωνεί απέλ, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την, ε, τις οδηγίες που αναφέρονται στην έκθεσή της ιδιαίτερα αυτή για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και μάλιστα με το σωστό τρόπο όλοι όσον αφορά ε, όντως υπάρχουν δύο χώρες το Λουξεμβούργο και η Ισπανία που καθυστερούν και η Κομισιόν προσέφυγε στο 10 τον Ιούνιο του 2008. Επίσης, οι οποιασδήποτε ε, εντάξει στις εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να γίνονται σωστά. Ε, προσφέραμε τη βοήθειά μας για να γίνει σωστή ε, ένταξη στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν έγινε κάτι τέτοιο και που ε, όπου ορισμένα πράγματα εναρμονίζονται με διαφορετικό τρόπο. Για αυτές τις περιπτώσεις Κομισιόν δεν θα να προσφύγει για παράβαση. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές τώρα πράγματι υπενθυμίζουμε ότι πλήρης εναρμόνιση για το θέμα αυτό ε, θεωρήθηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θα αποτύχανε συζητήθηκε το θέμα κατά τη έγινε διαβούλευση είχε γίνει πρόταση έγινε διαβούλευση έγιναν συζητήσεις στο Συμβούλιο και είδαμε ότι πραγματικά δεν είχε νόημα να ε, ευρύνουμε, διαβρύνουμε την οδηγία για να καλύψουμε και αθέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά τώρα επιθετικές πρακτικές που ρυθμίζονται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της οδηγίας UCP αυτές οι πρακτικές σχετίζονται μόνο με ε, σχέση καταναλωτή επιχείρησης δεν αναφέρονται στη σχέση επιχειρήσεων μεταξύ τους consumer protection legislation. Όσον από εκεί και πέρα η Κομισιόν θα συνεχίσει να προωθεί νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή μέσω του σχετικού δικτύου και θέλουμε πραγματικά τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για το SWIPS ως ε, ε, εργαλείο ανάπτυξης και το Κοινοβούλιο υπέβαλε σχετικό αίτημα και γι' αυτό η Κομισιόν ανταποκρίνεται και η δεύτερη εκδοχή του scoreboard των καταναλωτών θα δημοσιευθεί, θα είναι έτοιμη κατά τη διάρκεια του SWIPS. Από εκεί και πέρα για τις ε, εκστρατείες συνειδητοποίησης των καταναλωτών και τις σχετικές ιστοσελίδες και τα λοιπά και η, η Συμφωνία Απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα φτιάξει μια ιστοσελίδα το σελίδα με τίτλο Is It Fair για τον θεμητό ανταγωνισμό και τις θεμικές, θεμητές πρακτικές και ελπίζουμε να συνεργα... συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέμα τις εμπορικές πρακτικές και την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε φέτος και την εποπτεία της σωστής ένταξης εθνικές νομοθεσίες και της σωστής εφαρμογής. Ευχαριστώ. Και αυτή η έκθεση θα ψηφιστεί αύριο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να δηλώσω προς την κυρία Βάιλερ ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για τη διεκπαιρέωση της έκθεσης αυτής βασίζεται σε μια απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Πού προχώρησε για τη δικασία αυτή. Έχουμε τώρα την εξέταση της έκθεσης Γκερέιδο. Κοινή αλληλευτική πολιτική και προσέγγιση διαχείριση της αλληλείας με βάση το οικοσύστημα. Ο κύριος Γκερέιδο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ανακοίνωση βασίζεται